Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. εγκρίνονται τα πρακτικά, τα συνοπτικά πρακτικά. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της ε, Αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπά της εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας με θέμα Σουδάν και Νότιο Σουδάν. Δίνω το λόγο στον ε, κύριο ε, Βάμεν Νικολάη, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Υπάτης Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας. Έχετε το λόγο, κύριε Βάμεν. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ομιλώ εξ ονόματος ε, της είπα της εκπροσώπου Αντιπροέδρου Άστον, η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα εδώ για να συζητήσει την κατάσταση μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν που επιδεινώνεται διαρκώς. Πράγματι, με μεγάλη ανησυχία είμαστε μάρτυρες των αυξανόμενων εντάσσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Φτάσαμε σε μια κριτική περίοδο τον περασμένο μήνα με την κατάληψη και την κατοχή των ε, κοιτασμάτων πετρελαίου του Χέγλικ από τον Νότιο Σουδάν και τις συνεχιζόμενες ε, αεροπορικές επιθέσεις κατά της, επικρα... από επικράτειας του Νότιου Σουδάν από το Σουδάν. Η ΕΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος καταδίκασε δρυμύτατα τις ε, ενέργειες αυτές και των δύο πλευρών τις οποίες κάλεσε να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στο τραπέζι των τραυματεύσεων. Ο πρόεδρος Βαν Ρομπό τηλεφώνησε στον πρόεδρο του Νοτιού Σουδάν Σαλβακίρ και του ζήτησε να σταματήσει αμέσως και να προβεί αμέσως στην ε, απόσυρση των δυνάμεων. Το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων στις 23 Απριλίου χαιρέτησε την ε, απομάκρυνση του Νότιου Σουδάν από το Εγκλίγ μετά από έντονη ε, διεθνή πίεση και ζήτησε την κατάπαυση των εθνοπραξιών το ταχύτερο δυνατό. Στις 24 Απριλίου η Αφρικανική, το, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας θέσπισαν έναν οδικό χάρτη με μία σειρά από σαφή βήματα και χρονικά περιθώρια ώστε να τεθεί ένα τέρμα στις εχθροπραξίες ώστε και να επιστρέψουν στα τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά από αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ομόφωνα ε, ψήφισε το ψήφισμα 2046 της 2 Μαΐου που ενέκρινε και δέχθηκε τον οδικό χάρτη του, της Αφρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για σημαντικό βήμα. Τώρα όμως έχουν συνδυάσει, έχουν συνδυάσει τα λόγια με τις πράξεις. Πρέπει τα μέρη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενεργοποιήσουν την κοινή αποστολή επαλήθευσης και παρακολούθησης των συνόρων. Στη δήλωση της στις 5 Μαΐου η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος χαιρέτησε θερμά τον ε, οδικό χάρτη που περιέχεται στο ψήφισμα 2046 του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε και τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν αυτό το ψήφισμα χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Τα μέρη τώρα έχουν τρεις μήνες στη διάθεσή τους για να καταλήξουν στη συμφωνία για όλα τα θέματα που εκκρεμούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη θα προτείνουν συγκεκριμένε προτάσει για τη διευθέτηση τη διαφορά. Αν δεν υπάρξει μόρφωση, το Συμβούλιο Ασφαλεία έχει απειλήσει ότι θα επιβάλλει μη στρατιωτικέ κυρώσει. Ο δικός χάρης αναφέρεται επίσης και στη σύγκρουση στο Νότιο Κορντοφάν και τα κράτη του γαλανού Νείλου που συνδέονται με τις ε, τρέχουσες εντάσεις ανάμεσα στο Σουδάν και τον Νότιο Σουδάν. Η κυβέρνηση του Σουδάν πρέπει να επιτρέψει πρόσβαση, άμεση πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους ε, τον άμαχο πληθυσμό που, έχουν, που έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση. Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική διευθέτηση απαιτείται για την επίλυση της ε, διαφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλέσει την κυβέρνηση του Σουδάν και όλες τις ε, άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές να συμμορφωθούν με τα αιτήματα και τις ε, απαιτήσεις του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια εθνική μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και στις δύο χώρες είναι μια σημαντική ευκαιρία με την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται όλοι σε αυτή τη δικασία. Στο Βορρά ανησυχούμε πολύ για την, για την κράτηση ε, των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ε, πολιτικών της αντιπολίτευσης και απλών ειρηνικών φοιτητών που διαμαρτύρονται. Μια από τις βασικές αρχές της ε, ολοκληρωμένης ειρηνευτικής συμφωνίας ήταν η εγκαθίδρυση δημοκρατικής διακυβέρνησης με βάση την πολυμέρεια και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Στο Νότο κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης μας απασχολεί. Χαιρετήσαμε την πρόσφατη επίσκεψη του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβη Πιλάρη στο Νότιο Σουδάν με σκοπό να βοηθήσει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην έννοια των δύο βιώσιμων κρατών. Ε, ε, ευχαριστηθήκαμε όταν ο πρόεδρος Σαλβακύρη επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες τον Μάρτιο και μας ενημέρωσε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, συμφωνία, ε, εταιρική συμφωνία και στη σύμβαση του Κοτονού. Αυτό θα δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για μια μελλοντική αναπτυξιακή συνεργασία. Ω εταίροι μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για τα θέματα αυτά και για τι θεμελιώδει αρχέ αυτή τη εταιρική σχέση που είναι η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια για τον Νότιο Σουδάν με τη μορφή ειδικών κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο αναπτυξιακό ταμείο συνολικού ύφους 285 εκατομμυρίων ευρώ. Υποστηρίξουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης του Νοτιού Σουδάν και, του Σουδάν και τις, πρωτο, και τις ε, προσπάθειές του να ενισχύσει τους θεσμούς του, να υποστηρίξει την αγροτική ανάπτυξη και τη γεωργία, την υγεία και την παιδεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζει επίσης ε, διάφορες αποστολές για να αυξηθεί η ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τζούμπα για το Βορρά λυπούμαστε για την κυβερνητική απόφαση της μη επικύρωσης της Συμβασής του Κοτονού του 2005. Παρόλα τα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κονδύλια για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε περιοχές όπως τον Ταρφούρ, το Ανατολικό Σουδάν, το Νότιο Κορδοφάν και τον ε, Γαλανό Νίλο. Αυτή είναι μια προσθήκη στο ευρύτερο πρόγραμμά μας ανθρωπιστικής βοήθειας ε, Υπάρχουν όμως ακόμα 1,7 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που κατοικούν σε καταβλισμούς. Η κοινή ειρηνευτική αποστολή η UNAMID αντιμετωπίζει ακόμα περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεών της από την κυβέρνηση του Σουδάν. Χαιρετίζουμε το έγγραφο του Ισδόχα για ειρήνη στον Ταρφούρ σαν θετικό βήμα για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ειρηνευτικής διαφθέτησης των διαφορών που πρέπει ωστόσο να εφαρμοστεί πλήρως. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά επανάληψη έχει υπενθυμίσει την υποχρέωση της κυβέρνησης του Σουδάν να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σύμφωνα με το ψήφισμα 1593. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κατάσταση του Σουδάν και του Νότιο Σουδάν παραμένει ε, στοιχείο μεγάλης ανησυχίας. Κατέστα σαφές, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επανέλθει η ειρήνη και η σταθερότητα και στις δύο χώρες παραμένουμε προσιλωμένοι στην ανάγκη υποστήριξη της ανάδυσης δύο βιώσιμων κρατών σε συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης. Ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Χριστιανοδημοκρατών. Δίνω το λόγο στον κύριο Μίτσελ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και το Συμβούλιο για την πρωινή παρουσίαση που μας έκανε και, το, και την απογευματινή παρουσία. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Ε, αναφέρεται ότι η χώρα αυτή έχει καταστραφεί από βιοπραγίες που συνεχίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό και σκεφτήκαμε ότι η απόσχηση του Νοτιού Σουδάν θα οδηγήσει τουλάχιστον ε, σε μία εξομάλυση της κατάστασης προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Οι άνθρωποι δυνοπαθούν, υπάρχουν πολύ εκτοπισμένοι. Εκτός ότι έχουμε μία περιοχή με πλούσια ορυκτά κοιτάσματα και πλούτο. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να αναχαιτήσουμε κάπως ε, την όξυνσή της και να αντιμετωπίσουμε την δυνότατη ανθρωπιστική κρίση, ιδιαίτερα στους καταβλισμούς προσφύγων εκτός του Σουδάν, ο κόσμος συνοστίζεται. Θα πρέπει εκεί να εξασφαλίσουμε υποστήριξη και εφόδια για τους ανθρώπους αυτούς, ε, ώστε να υπάρξει μια προστασία και ασφάλειά τους. Τώρα, η κατάσταση μεταξύ Βορείου και Νοτιού Σουδάν είναι χαρακτηριστική περίπτωση του τι μπορεί να συμβεί μετά από απόσχηση όταν δεν υπάρχει σταθερότητα. Γιατί γιορτάζουμε την Αραβική Άνοιξη, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η, η επόμενη μέρα, γιατί πολλές από τις χώρες αυτές δεν έχουν τέτοια παράδοση διακυβέρνησης. Και συνεργαζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση και για κατάρτιση και για παροχή τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να αναπτύξουν το δυναμικό του και να μετατρέψουν την περιοχή του ε, σε σταθερή περιοχή. Δεν μπορούμε ούτε εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο ΙΕ να κάνει τα πάντα. Και υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα με μεγάλο κόστο και σε ανθρώπινε ζωέ και σε καταστροφέ αλλά σε τέτοιες περιοχές που οι άνθρωποι ε, εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τις εξαγωγές και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, η κατάσταση έχει το κόστος. Γιατί δεν μπορούμε σε νωρίτερη φάση να βρούμε αυτά τα κονδύλια ώστε να επενδύσουμε με την Αφρικανική Ένωση και να εξασφαλίσουμε ε, ανεφοδιασμό αυτών των ε, κρατών και καλύτερη διακυβέρνηση ώστε να αποφεύγουμε όξυση των κρίσεων. Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τεράστιες προσπάθειες για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Και πραγματικά έχει δαψιλώς χρηματοδοτήσει την πρόσβαση του Νοτιού Σουδάν στην ανεξαρτησία. Ε, στηρίζοντας την ε, συμφωνία την ειρηνευτική του 2005 γιατί ήταν ή η συμφωνία αυτή ή ο πόλεμος. Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Το πρόβλημα τότε δεν είχε ακόμη επιληθεί. Κανένα πρόβλημα δεν είχε διαθετηθεί. Ούτε το θέμα της ηθαγένειας, ούτε το νόμισμα, ούτε το θέμα του χρέους και ούτε πάνω απ' όλα το θέμα της κατανομής ε, των ε, κοιτασμάτων πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, του Σουδάν και του Νοτιού Σουδάν. Και μας έχει έρθει ως μπούμερανγκ αυτή η μη διαθέτηση των προβλημάτων. Και το χειρότερο είναι ότι εδώ και ένα χρόνο έχουμε την Κίνα που σε διεθνές επίπεδο, ακριβώς επειδή ελέγχει όλη την αλυσίδα του πετρελαίου από την ε, εκμετάλλευση μέχρι τα δηληστήρια και αγοράζει το πετρέλαιο, ξαφνικά θα λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έκανε τόσα πολλά ξαφνικά έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο και είναι ενοχλητική αυτή η κατάσταση. Χαιρετίζω το άρθρο 4066 του ΙΕ που είναι ένα τεράστιο βήμα πρόοδου και συμφωνούμε και θα ήθελα να εκφράσω τρεις επιθυμίες. Η πρώτη επιθυμία είναι επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει αποστολές παρατήρηση εκλογών γιατί γνωρίζαμε ότι είναι έθραυστη αυτή η χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα follow-up, μια συνέχιση μετά την παρακολούθηση, την παρατήρηση των εκλογών και στο Σουδάν. Επίσης, προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κάνει τόσα πολλά Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχει πασχίσει για τις χώρες αυτές και συνεχίζει μέσω και της της εκπροσώπου. Θα πρέπει η φωνή της να γίνει ακουστή γενικώ. Επίσης θα ήθελα η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μια ισορροπημένη θέση μεταξύ του Βορείου και του Νότου να ε, να αναφερθεί πέρα του ICC και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή και τη θέση του, του πρόεδρου Μπασίρ. Επίσης, ό,τι αφορά τις πολιτείες Blue Nile και Νότιο Κορδοφάν, ε, η κατάσταση είναι πραγματικά αν, άνω ποταμών. Δεν έχουμε εξασφαλίσει μέχρι στιγμής πρόσβαση στις περιοχές αυτές. Ε, περιοχές που καθημερινά αντιμετωπίζουν μια ανθρώπινη τραγωδία. Ευχαριστώ της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ο κύριος Σαρλ ε, Γκέρνς, για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέραν της προσοχής που χρήζει αυτή η διαμάχη μεταξύ Βορείου και Νοτιού Σουδάν, ε, έχω και προσωπικό ενδιαφέρον γιατί ήμουν ε, ένας από τους υπογράφοντες της ε, Γενική Ειρηνευτικής Συμφωνία του 2005 στο Ναϊρόμπι και εκεί έβαλα την υπογραφή μου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι κάτι πρωτοφανέ. Ήταν γνωστό και πριν από την ανακήρυξη τη ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν και ακόμη και, μετά, και στην υπογραφή τη συμφωνία πέντε χρόνια μετά τότε όλοι αναγνωρίζαμε ότι δεν χωρεί εδώ στρατιωτική λύση στη διαμάχη, αλλά έχουν αλλάξει διαστάσεις. Μετά την ανεξάρτηση του Νοτιού Σουδάν δεν είναι ε, μια διαμάχη μεταξύ ε, δύο κομμάτων στην ίδια χώρα, αλλά έχει μετατραπεί σε διεθνή διαμάχη. Οπότε θα πρέπει να ισχύσει εδώ το διεθνές δίκαιο και οι λύσεις να αναζητηθούν σε επίπεδο διεθνούς ε, δικαίου. Θα ήθελα να ε, επενέσω εδώ τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που, έκαναν, που έκανα ό,τι μπορούσε. Θέλουμε να ε, βρεθεί μια λύση που θα τηρεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου και επίσης θα πρέπει για να διαθετηθεί αυτή η σύγκρουση, να εξαντληθούν όλα τα μέσα που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Μετά τις πολλαπλές προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αφρικανικής Ένωσης και μετά το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της ε, Αφρικανικής Ένωσης και μετά το ψήφισμα 2046, ε, είναι γνωστά τα σημεία αναφοράς για την ειρηνευτική διαδικασία. Και οι προσπάθειες των Αφρικανικών φορέων είναι πολύ χρήσιμες και τις υποστηρίξαμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή του 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και σήμερα είναι ένας απαραίτητος εταίρος των δύο χωρών ε, που προέκυψε μετά από τη, το, του Σουδάν. Είμαστε οι πρώτοι σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας, σε αναπτυξιακή βοήθεια, στη, στον ειρηνευτικό διάλογο, κατέχουμε ένα από τα κλειδιά της λύσης για την κατάσταση. Ένα από τα κλειδιά, αλλά όχι το μοναδικό κλειδί. Γιατί ένα από τα αίτια της αιτία ε, της διαμάχης είναι η φτώχεια, η εξαθλίωση που υπονομεύει τις βάσεις οποιασδήποτε βιώσιμη σταθερότητα Και το Νότιο Σουδάν και το Βόρειο Σουδάν είναι συνυπεύθυνοι για να ανέβρουν μια λύση. Θα πρέπει να σταθούν αντάξει των περιστάσεων δεν αρκεί να έχει κανεί ένα κράτο. θα πρέπει να μπορεί να το διακυβερνά κιόλα. Θα πρέπει να βρεθούν λύσει, γιατί αν δεν βρεθεί η λύση θα επανέλθουμε στην σύγκρουση και μέχρι σε 10 χρόνια είχαμε 2 εκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ χάθηκαν. Ελεύθερη ε, Συμμαχία, η συνάδελφος κυρία Γιούντιθ ε, Σαρτζεντίνη για λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από το Συμβούλιο και έχω έτσι μια, νιώθω μια ανασφάλεια. Όλοι προσπαθούν κατά την άποψή μου να μπουν στα φώτα της δημοσιότητας. Πρέπει όμως να σας πω ότι όλοι μας ε, λόγω της ε, κατάστασης στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν, μα όλοι μας ε, φέρουμε ευθύνη. Βεβαίως χαιρετίζω και εγώ το γεγονός ότι το Συμβούλιο ασφαλείας καθορίζει ή ενέκρινε το χάρτη πορείας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα το Νότιο Σουδάν δέχτηκε να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Αμπύρ αλλά ας δούμε λιγάκι πως έχει τώρα η κατάσταση νοτιο σουδαν δεχτηκε να αποσυρει τις δυναμεις του απο το αμπιρ ότι ε, θα έχουμε μια σύγκρουση που μπορεί να, συγκρου... συγκριθεί με τη σύγκρουση ανάμεσα στην Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Θα είναι μια σύγκρουση που θα έρχεται και επανέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν τη συγκρίνω με τη σύγκρουση Ερυθρέας-Αιθιοπίας. Πραγματικά φοβάμαι ότι και οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν τη συνοριακή σύγκρουση για να μην κάνουν τίποτα, για να αφήσουν να βασιλεύει η πείνα και η εξαθλίωση. Στο Νότιο Σουδάν θα αρχίσουν σύντομα οι βροχές. Απο, αποτέλεσμα αυτού το 60% της χώρας θα είναι παντελώς απροσπέλαστο. Ε, δεν θα μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιήσει τους δρόμους λόγω των βροχών. Τα αποθέματα τροφίμων για τον πληθυσμό μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί. Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε για χαρτιπορίες, για ειρνευτική διαδικασία, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μεριμνήσουμε να έχουν οι άνθρωποι ε, επαρκή τρόφιμα. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Το Νότιο Σουδάν δεν είναι σε θέληση να εξασφαλίσει μέλλον για τους πολίτες του. Και αυτό οφείλεται στο ότι το Νότιο Σουδάν δεν πουλάει πλέον πετρέλαιο. Κατανοώ τι σημαίνει αυτό, αλλά αν το Νότιο Σουδάν δεν μπορεί πλέον να φροντίσει για τους ε, κατοίκους του, τότε τι συμβαίνει. Τι είναι πιο σημαντικό, η σύγκρουση με τους γείτονες ή η ε, παροχή τροφίμων στους ε, κατοίκους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, το Νότιο Σουδάν να μπορεί πάλι να λειτουργήσει και να βρει αγορά για το πετρελό του. Ευχαριστώ. και Μεταρρυθμιστών είναι ο συνάδελφος κύριος Άνταμ Μπίλεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαμάχη του Σουδάν εδώ και χρόνια αποσπά την προσοχή του κόσμου. Αυτή τη στιγμή ε, και μετά την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν δεν έχουμε πια εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε πια τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς διαμάχης και επιπλέον αν ο στρατός του Νότου υποστηριχθεί από το στρατό της Ουγκάντας ίσως έχουμε μια περιφερειακή ανάπλη διαμάχη. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της διεθνούς κοινότητας απέναντι και στα διαιτήματα του Σουδάν ίσως φαίνονται ακατανόητες ο Νότος προσπαθεί να ε, υλοποιήσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και ε, απέσυρε τη, τη στρατεύματα από την επίμαχη περιοχή Χέγκλιγκ αλλά ε, ο κόσμος παρόλο που επίσημα στυλιτεύει τις δράσεις της κυβέρνησης του Χαρτούμ δεν αναλαμβάνει κυρώσεις εναντίον της. Επίσης δεν υπάρχει μια συστηματική στρατηγική για να αντιμετωπίσει αναθέτουν τα προβλήματα των προσφύγων, να έχουμε ε, ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ ανθεί το λαθρεμπόριο όπλων με τη συμμετοχή Κίνας, Ρωσίας, Λευκορωσίας ε, και θα πρέπει να καταδικαστεί αυτό το λαθρεμπόριο όπλων. Πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες του Νοτιού Σουδάν που παραμένουν ε, σε παραμεθόριες περιοχές μεταξύ Βορράς και Ρώτου δεν έχουν ρυθμισμένο ε, νομικό καθεστώς. Συνεχίζονται οι εθνοκαρθάσεις και μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μέχρι στιγμή δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο ελεύθερης διακίνηση στην παραμεθόρια περιοχή και ίσως χρειαστεί χάραξη των συνόρων σε ορισμένε περιοχές, νέα χάραξη των συνόρων. Ε, για να γίνει πιο αυστηρή η πολιτική του, της απέναντι στο Χαρτούμ θα αρκούσε απλώς ε, η, η δίωξη του Μπασίρ και η κατηγορία του από το Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν θα πρέπει ε, η βιομηχανία του Πεδρελαίου και τα, τα ωφέλη από εκεί να γίνουν παραπέτασμα για να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή. Χρειαζόμαστε επικοδομητικές συνομιλίες και καλό την είπατε πρόσωπο να συμμετέχει ε, δραστηρία σε τέτοιου είδους συνομιλίες για τις παραμεθορές περιοχές. Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο συνάδελφος κύριος Μπάστιαν Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία έκθεση από την εμπόλεμη περιοχή Νούμα είναι πραγματικά απογοητευτικές. Εδώ και μήνες αυτή η περιοχή έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των νοτιοσυνδανικών αρχών. Προσπαθεί οι κάτοικοι να επιβιώσουν όπως μπορούν στις ορεινές περιοχές. Μεγάλος αριθμός ε, προσφύγων βρίσκεται στη, στον καταβλισμό στο Νότιο Σουδάν. Αρκεί να διαβάσει ε, κανεί την εσωτερική έκθεση τη Παγκόσμια Τράπεζα που απροκάλυπτα μιλά για δραματικέ συνθήκε. Το ανεξάρτητο Νότιο Σουδάν, στο ανεξάρτητο Νότιο Σουδάν. Πρέπει, τι, πρέπει λοιπόν να δοθεί βοήθεια σε αυτές τις χώρες αλλά μια ανεύθυνη, μια ανεύθυνη συμπεριφορά ανίκανων, ανίκανων ε, πολιτικών υπό την προεδρία του Προέδρου Σαβακύρ. Τα έσοδα του κράτους και ο νεποτισμός και η διαφθορά αποδεικνύουν αυτή την θρυβερή διαπίστωση. Υψηλό ποσοστό των Νότιων Σουδανών έχουν ξεπεράσει το όριο της φτώχειας και το 2013 πιστεύουμε ότι θα φτάσει το ποσοστό στα 83% το 2013. Ε, απευθύνομαι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δωρητές θα δώσουν, θα δώσουν μια σαφή προειδοποίηση στον πρόεδρο αυτό. της ε, Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων χωρών, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Σαμπίνε Λέουζινγκ Για δύο λεπτά. Πάλι λοιπόν πόλεμος για το πετρέλαιο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς ε, να χαρακτηρίσει τα γεγονότα στο Σουδάν. Και ο άμοχος πληθυσμός και των δύο χωρών υποφέρει τα μάλα. Ε, είναι σαφές ότι όλες οι πράξεις βίας πρέπει να καταδικαστούν. Οφείλουμε να αναζητήσουμε μια ειρηνική λύση των ε, συγκρούσεων. Αυτό όμως δεν μας δεσμεύει ε, στο να μιλάμε για τα αίτια και να ρωτάμε το κατά πόσον μια καλύτερη και μεγαλύτερη στράτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόσπαση του Νότιου Σουδάν ήταν σωστή ή όχι λόγω των καταστάσεων που ακολούθησαν. Σίγουρα δεν υπάρχει ασφαλής λύση, όμως είναι εξίσου σαφές ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με βία. του αντίον είναι απολύτως απαραίτητα να ε, διατηρηθεί το εμπάργκο όπλων για να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι από το 2004 υπάρχει εμπάργκο ε, παράδοσης όπλων απέναντι στο Σουδάν και από το 2011 ισχύει το εμπάργκο αυτό και κατά του έναντι του Νοτίου Σουδάν. Ε, τότε ελέγχθη ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις στο Νότιο Κάτι το οποίο δεν έγινε. Όσο και αν είναι δύσκολο, οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις πρέπει να επιταθούν. Αν η διεθνής κοινότητα θέλει να παρέμβει ε, θετικά, τότε αυτό μπορεί να το πράξει μόνο με το ρόλο ενός ουδέτερου διαπραγματευτή και χωρίς να εκφράζει αυτό συμφέροντα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν ουδέτερος και γι' αυτό ανησυχώ κατά πόσον τέτοιου είδου σενάρια μπορούν να έχουν μέλλον. Και φοβάμαι ότι θα υπάρξουν και άλλες περιοχές πλούσιες με πετρέλαιο ε, στην Νότια Αφρική που θα αποσπαστούν και αυτές. Ε, το ε, στοιχείο, το εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής ε, και η δημιουργία κρατών δεν μπορεί να είναι η λύση. Ούτε είναι σωστό να παρεμβαίνουμε ε, στα εσωτερικά κρατών ε, γιατί αυτό δεν επιφέρει ειρήνη αλλά θάνατο και εξαθλίωση. Συνάδελφος κύριος Ανδρέας για 1,5 λεπτό. Στο Σουδάν αγωνίζονται για να αποτινάξουν το ζυγό των απεικιοκρατών. Ε, στο Βορρά υπάρχουν ε, συνεχώς ε, διαμάχες ανάμεσα στις εθνότητες για το νερό, γίνονται βιασμοί, όλα αυτά κλιμακώνονται πολύ εύκολα στο Σουδάν. Σε αυτή τη χώρα έχουμε πολλές γενιές που μεγάλωσαν χωρίς τα βασικά αγαθά και χωρίς να υπάρχει υποδομή ότι λέγεται τη μία μέρα, την άλλη μέρα δεν ισχύει. Κατόπιν τούτου οι ειρηνευτικέ συνομιλίε δεν είναι εύκολε. Ο ειδικό απεσταλμένο τη Αφρικανική Ένωση, ακόμα και αν καταφέρει να, επανε, ε, να επιτύχει την επανέναρξη των συζητήσεων, παρόλα αυτά η κατάσταση θα είναι ευαίσθητη. Και ακόμα και αν εξευρεθεί ε, ειρηνική λύση, παραμένει ένα τεράστιο δυναμικό σύγκρουση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να επανέλθει ε, επανέλθουν τα βασικά αγαθά, μακροπρόθεσμα. Δεν φτάνει το πετρέλαιο της ε, χώρας για να ε, επανεκκινηθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού. Η βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, πρέπει ε, να εκφράζει και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Με βάση το κινέζικο μοντέλο θα μπορούσε κανεί την ανθρωπιστική βοήθεια να τη συνδέσει με το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει πετρέλαιο στο Βόρειο Σουντάν και τα αποθέματα αυτά μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Ε, όσον αφορά τα κοινοτικά, τα δικά μας κονδύλια για το Σουδάν, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παράνομη μετανάστευση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επεξεργαστούμε και μια συμφωνία επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών. Είμαστε στην ενότητα άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές. Πρώτη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Μαρίγια Ντελτσεβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σχέση μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν όλο και χειροτερεύουν. Ανησυχούμε βλέποντα την υποβάθμιση τη κατάσταση τη ανθρωπιστική και τη ασφάλεια στην περιοχή. Ένα χάρτη πορεία εγκρίθηκε και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Αλλά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμή ε, δεν είναι επαρκή διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι βομβερδισμοί και άλλες στρατιωτικές επιθέσεις από πλευρά του δανεικού στρατού. Η ανθρωπιστική κατάσταση των αμάχων επιδεινώνεται και οδηγεί σε εκτεταμένες μετακινήσεις ατόμων το θέμα επίγει. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες και ένα χρονοδιάγραμμα που θα συμβάλλει στην πρόθεση της διαδικασίας. Η πρώτη συνάντηση του κοινού μηχανισμού για τα πολιτικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό ώστε οι προτεραιότητες ασφάλειας και δρέως της ειρήνης να εντοπιστούν και να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης. Ε, ε, το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή των διεθνών εταίρων που πρέπει να δεσμευθούν για να στηρίξουν τις προσπάθειες των δύο δύο πλευρών και η, ένας, η δημιουργία ενός ε, κοινού μηχανισμού ελέγχου των συνόρων είναι σημαντικό στοιχείο για τη διεθνή δράση που πρέπει να αποτελέσει εγγυήσει ώστε οι αποφάσει θα ληφθούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Αφρικανική Ένωση πρέπει να συνεργαστούν στενά μεταξύ του και να υλοποιήσουν τι υποχρεώσει του, αναλαμβάνοντα πλήρω το ρόλο του εταίρου. Να έχουν δηλαδή το θάρρο επίση να θέσουν το θέμα των κυρώσεων. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, να, μεγαλύτερη δραστηριότητα για την, ε, ε, για, την ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί να στέλνουμε απεσταλμένους για τον έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας και να μην παρέμβουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να μετατρέψουμε τις, τα λόγια σε πράξη. Ο ρυθμός σας υπάρχει πρόβλημα στη διερμηνία. Είστε χυμαρόδης. Je finis, le Président, et je les interprètes nous devons faire preuve de courage pour que les textes puissent se transformer en actes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Την ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Να καταβάλουμε όλε τι προσπάθειε για την ειρηνευτική επίληψη αυτή τη σύγκρουση και να δώσουμε όλη την απαιτούμενη στήριξη στου πολίτε των δύο χωρών. Ε, καλώ στο βήμα την κυρία Άννα Γκόμε για ένα λεπτό περίπου ένα χρόνο μετά την ανακήρυξη της ε, ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν, όπως είχαμε προβλέψει πολύ, οξύθηκαν οι σχέσει μεταξύ των δύο πλευρών με βιοπραγίε, αντίπεινα, όξυση των εκκρεμών θεμάτων όπως η κατανομή των πετρελαίων και ε, κοιτασμάτων, ε, την κατάσταση του ABA και η διαθέτηση των παραμεθόριων περιοχών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δέσμευση τουλάχιστον στην εφαρμογή του οδικού χάρτη για να ε, σταματήσουν οι εχθροπραξίες ε, και αυτό με την υποστήριξη ε, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Αφρικανικής Ένωσης. Και επίσης θα πρέπει να απαιτήσουμε παράδοση του Πρόεδρου Μάναρ Βασίλη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να συνεχίσουμε με την παρατήρηση των εκλογών. Αυτή είναι η στόχη για, τον εκδημοκρατισμό και του Νοτιού Σουδάν. Το έργο της ΥΠΑ της εκπροσώπου θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες να αποκτασταθεί το δυναμικό διακυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν. Αλλιώ δεν πρόκειται να έχουμε βιώσιμε ειρηνευτικέ διαδικασίε για την περιοχή. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει ε, δεόντω το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων ε, στην περιοχή αυτή που αντιμετωπίζουν τεράστιε δυσκολίε προσπαθώντα να βοηθήσουν του χιλιάδε εκτοπισμένου και θύματα τη διαμάχη. Είναι ο συνάδελφο κύριο Νικολό για λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Νότιο Σουντάν ε, δεν είναι πλέον αυτή η ευχάριστη είδηση που είχαμε πριν από ένα χρόνο. Οι πολίτες ε, τόσο του Σουδάν όσο και του Νότιου Σουδάν δεν γνωρίζουν ούτε την ειρήνη ούτε τη σταθερότητα πόσο μάλλον ανάπτυξη. Περπατάνε με τα πόδια, μεγάλες αποστάσεις διασχίζουν για να βρουν νερό. Αυτό μας λέει κάποιος που γνωρίζει την περιοχή ε, και σήμερα μας λένε επίσης ότι πολλές φορές όταν περπατάνε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να τυναχτούν στον αέρα από κρυμμένη νάρκη και νερό δεν βρίσκουν και πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο να πάει κανείς στην Τζούμπα ούτε στο Καρτούμ. Νομίζω ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις μελέτες της πρέπει να βασίζεται σε εξής αρχές. Πρώτον να κρατήσει ζωντανή την προσοχή προς αυτή την περιοχή. Να μην υπάρχει κίνδυνος η κρίση να ξεχαστεί, να είναι κάτι το οποίο βάλαμε στο θεματολόγιο, το βάλαμε σε ένα ντουλάπι και δεν ασχολείται πλέον κανείς ούτε τα μέσα ενημέρωσης ούτε η διεθνής κοινότητα. Πρέπει να επιμείνουμε στο να εφαρμοστεί το 20 46 ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για αυτά που συμβαίνουν στο Καρτούμ. Γιατί ο πρώην πρόεδρος του ε, Σουδάν είπε ότι περιμένει ε, στο Σουδάν να γίνουν αυτά που έγιναν ε, γενικά με την Αραβική Άνοιξη. Έχει αποτύχει η διοίκηση και ο Μπασίρ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι και να μην επαναληφθεί αυτό το οποίο έγινε στη Βόρεια Αφρική. Τέταρτο σημείο της παρέμβασής μου. Εμείς είμαστε βασικοί δωρητές στο Νότιο Σουδάν και πρέπει πρέπει να εφαρμόζεται καλύτερα ο νόμος στην στη Τζούμπα. Σήμερα ε, αυθαίρετα κάνει κανείς ό,τι θέλει. Πρέπει λοιπόν να επανέλθει η αξιοπιστία των κομμάτων στα μάτια των πολιτών και αυτό είναι πολύ δύσκολο αν δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποιο αποτελεσματικό δικαστικό ανεξάρτητο σύστημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελειώνω γρήγορα και με ένα άλλο σημείο επί το οποίο είχαμε πιστεί στην προσοχή, δηλαδή ε, για το Νότιο Σουδάν να υπάρχει υπάρχει ένας, ένα ταμείο διαφανές που να συγκεντρώνει ε, τα έσοδα από το πετρέλαιο. Όπως συμβαίνει και στο Τιμόρ. Το Τιμόρ είναι μια πολύ καλή και θέλω αυτό να συμβεί και στο Νότιο Σουδάν. Είναι ο συνάδελφος ε, κύριος Φιωρέλο Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ελέγχθησαν σχετικά με το επίμαχο θέμα των ε, εκτάσεων των εδαφών ε, και του πετρελαίου. Η συνέπεια ήταν ότι τα κράτη συμφώνησαν να ε, διαχωριστούν. Η γενική κοινότητα παρακολουθεί πλέον να υπάρχει μια ένοπλη σύραξη στην περιοχή αυτή. Ένα άλλο ε, τραγικό γεγονός είναι ότι το Σουδάν μπλοκάρει ανθρωπιστική βοήθεια που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, περίπου 200.000. Η Ευρώπη πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια θα ήθελα να εφαρμόζει μια πιο στρατευμένη πολιτική ε, απέναντι στην Αφρικανική Ένωση και όχι μόνο με ε, κινέζικη επιρροή ή επειδή υπάρχει κινέζικη επιρροή αλλά κυρίως για να δοθεί σημασία στην παναφρικανική πολιτική και έτσι ώστε η Αφρική να ανήκει περισσότερο στους ίδιους Αφρικανούς. Ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος ε, του, ε, οικονομικού, της οικονομικής νεοαπικιοκρατίας σε αυτή την περιοχή. Ε, ακολουθεί στο βήμα ο συνάδελφος κύριος Βίλι Μέγερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Λέσσινγκ, η συνάδελφος, σας παρουσίασε τη θέση της ομάδας για την σύγκρουση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να αυταπατώμαστε. Όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε του Ισραήλ και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξαν και χρηματοδότησαν την απόσχηση του Νοτιού Σουδάν χωρί να έχουν ε, επιλύσει προηγουμένω ε, τα εκρεμή θέματα ε, για τα 2.000 χιλιόμετρα και η μεταφορά του αργού πετρελαίου γνωρίζουμε προς που βαδίζαμε. Τώρα διαρριγνύουμε τα ημάτια μας και εκπλησόμαστε για την σύγκρουση αυτή. Ουσιαστικά τη στηρίξαμε αυτή τη διαμάχη. Γιατί επρόκειτο για μια γεωστρατηγική δράση της δύση με μοναδικό στόχο να αποσυρθεί από τον αραβικό έλεγχο η πιο πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου περιοχή του Σουδάν για να ευνοηθούν ήδη. Όπως πάντα έχουμε την περίπτωση δύση και πετρελαίου. Και ενδιαφερόμαστε για την φτώχεια. Ποια είναι η σημασία που δίνουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας στη Δύση. Άλλο ένα πάθημα που θα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Γιατί πέραν των ε, ζητημάτων των ε, πετρελαϊκών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η φτώχεια και ο κόσμος που υποφέρει. Θεωρία είναι έμπλεα γεμάτα από επισκέπτες ε, και τους απευθύνω θερμό χαιρετισμό και εύχομαι ευχάριστη και παραγωγική διαμονή εδώ στο όμορφο Στρασβούργο. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Φίλιπ Κάτσμαρεκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, η ανακήρυξη ε, τη ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν στι 9 Ιουλίου του 2011 ήταν μια στιγμή χαρά και εκπλήρωση. Μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε μια νέα εποχή. Φαινόταν ότι οι προοπτικέ ε, του νέου κράτου ήταν καλή. Σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου που θα εξασφάλιζαν ε, καλό εισόδημα εθνικό. Ε, επίσης είχαμε ε, για τον Νότιο Σουδάν τη βοήθεια των ξένων δωρητών που το 2011 έδωσαν, ε, δήλωσαν βοήθεια 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρ' όλα αυτά μετά από λιγότερο από ένα χρόνο εξαρτησίας οι προοπτικές δεν είναι πια και τόσο ρόδινες. Γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε καλά το υπόβαθρο των γεγονότων. Στο Σουδάν δεν υπάρχει ουσιαστικά φορολογικό σύστημα. Θεωρητικά παρακρατούνται οι φόροι, αλλά στην πράξη το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Ακριβώς γι' αυτό τα έσοδα από την τις πωλήσει πετρελαίου ανέρχονται σε 97% του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχει βέβαια πρόβλημα γιατί το πετρέλαιο του Νοτιού Σουδάν μπορεί να μεταφερθεί στο λιμάνι του Σουδάν μόνο με ένα πετρελαγό που περνάει από το Σουδάν. Και είναι δύσκολο μέχρι πρώτη ως εχθροί να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γι' αυτό και υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ε, φαίνεται ότι το Νότιο Σουδάν προτιμά να μεταφέρει το πετρέλαιο μέσω της Κένιας προς τη Μομπάσα. Το Δεκέμβριο του 2011 συνήθη μια αρχική συμφωνία για τη δημιουργία νέου πετρελαγωγού. Βέβαια, ένα μήνα αργότερα, ο πρόεδρος Μπασίρ ε, έκλεισε το φόρο πετρελαγωγό, ε, κάτι που προκάλεσε τη διαμαρτυρία των Νοτιοσουδανών. Χωρίς διευθέτηση ε, του ζητήματος μεταφοράς του πετρελαίου δεν πρόκειται να εξασφαλίσουμε σταθεροποίηση της περιοχής. Κάτσμαρεκ, δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Αρλάτσι και επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Μαριέλε Ντεσαρνέζ για δύο λεπτά. Μάικρο. Vous m'entendez Oui, ça y η νέα δημοκρατία του Νότιου Σιδάν υπάρχει εδώ και δέκα μήνες, αλλά εδώ και πολλούς μήνες βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τον γείτονά της του Βορρά. Έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στα σύνορα και οι δύο αυτές χώρες που έχουν τα πάντα για να ανθίσουν και να αναπτυχθούν κατασπαταλούν τις δυνάμεις τους σε αυτό τον πόλεμο, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί τέτοιοι πόλεμοι πρέπει λοιπόν να τηρήσουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να ξεκινήσουν και πάλι τι διαπραγματεύσει ανεφόρων. Οι δύο νέε χώρε είχαν δεσμευθεί να το κάνουν αυτό, να ρυθμίσουν τα προβλήματά τους, να οριοθετήσουν τα σύνορά τους, το καθεστώ εκείνο που κατοικούν στο βορρά και το νότο και να μοιραστούν τα κοιτάσματα πετρελαίου ο Νότος έχει 70% των κοιτασμάτων, έχει κάθε συμφέρον να επιτύχει μια συμφωνία που θα ε, ε, ωφελήσει αμοιβαία και τις δύο πλευρές. Καμία χώρα δεν πρέπει να στηριχθεί στη σιωπή της ε, παγκόσμιας κοινότητας ενώπιον του ανθρωπιστικού δράματος που υπάρχει στη χώρα. Εάν δεν εισέλθουν, στο, αν δεν εισέλθουν μεταχέως στο Ντούμπα ή στο Νταρφούρ θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Η Κίνα έχει αναλάβει τις ευθύνες της Πολύ καλά. Αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προβάλλει την πολιτική της παρουσία και τη θέση της. Η ισόρροπη στάση μας είναι η καλύτερη. Ας την παρουσιάσουμε με μεγαλύτερη έμφαση και με, μεγαλύτερη ορατότητα και ας μην ξεχνάμε το, τη σύγκρουση και το δράμα στον Ταρφούρ. Επόμενος αγορητής είναι ο συνάδελφος κύριος Νικόλαος Σαλαβράκος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτυχία των μέχρι τώρα προσπαθειών για την ειρήνευση στα δύο ε, σουδανικά κράτη, ειδικά η αποτυχία της πρόσφατης ειρηνευτικής συμφωνίας, δεν αποτελεί καλό ιονό για τις πιθανότητες αποφυγής νέων συγκρούσεων που κρατάνε εδώ και δεκαετίες και συνεχίζουν την εξαθλίωση των δύο χωρών. Οι δύο χώρες είναι αλληλοεξαρτώμενες οικονομικά και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι συνεργασίας. Προς αυτόν τον σκοπό πρέπει να πάψουν τα δύο κράτη να υποθάλπουν και να στηρίζουν τους εχθρούς της άλλης πλευράς καθώς κάτι τέτοιο δυσχεραίνει την ειρηνευτική διαδικασία. η αποδυνάμωση του σουδάν λόγω της εξάρτησής του πλέον από τον νότο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των σχέσεων της χώρας αυτής με τους αφρικανούς γείτονες και αναμένεται να ενισχυθούν οι σχέσεις με αραβικές και ισλαμικές χώρες και με την άνοδο των ισλαμικών δυνάμεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό η οικονομική κατάσταση του σουδάν έχει χειροτερέψει αισθητά μέσα στο 2012 λόγω της πάυσης της ροής του πετρελαίου και έτσι αναμένεται η οικονομία να υποχωρήσει κατά 9,4% φέτος. εκτιμάται επίσης ότι ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 19% μέσα στο 2012 με ανωδικές τάσεις. Οι ενισχυτικές αυτές διαστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πράξει η ύπατος αρμοστία τα αδέοντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βράκο. Ε, ακολουθεί στο βήμα ο κύριος Κρίστιαν Ντάν Πρέντα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να καταδικάσω τους βομβαρδισμούς στο Βορρά, στο στο βόρειο τμήμα του Νότιου Σουδάν που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη βομβαρδισμοί του Βορείου Σουδάν. Σκέφτηκα αρχικά ότι δεν ήταν ενημερωμένα τα στοιχεία, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια νέα πρόκληση από πλευρά του Σουδάν. Κάτι που μας ε, ξοκάρει όλους κάτι που συμβαίνει λίγες μέρες ε, που ανακοινώθηκε ότι οι ηγέτες των δύο κρατών δέχθηκαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτές οι επιθέσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ε, δεν είναι διατεθειμένο το Σουδάν να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο Αλμπασίρ δεν φαίνεται να θέλει πραγματικά να διαπραγματευτεί τον χάρτη πορείας. Γι' αυτό καλώ τους διαπραγματευτές της Αφρικανικής Ένωσης και την ομάδα τους να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις και να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και ένας νέος πόλεμος στην περιοχή. Τέλος, θέλω να χαιρετήσω τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών για τις προσπάθειές να τηρήσουν την ειρήνη στην περιοχή. Η εντολή τους που έληξε χθε θα διευρυνθεί, θα επεκταθεί ώστε να ε, είναι πιο αποτελεσματικές και θα χρειαστεί επίσης να ενισχυθούν στρατιωτικές δυνάμεις. Μιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος ε, Γιάρος Βαλέσα για λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το Νότιο Σουδάν που μετά από πολύχρονη μάχη στην σύγχρονη Αφρική ε, αποσχίστηκε από το Βόρειο Σουδάν ε, δεν έχει εξασφαλίσει μια ευήμερη διαβίωση. Μετά από την τραγική ιστορία έχει περάσει μια κατάσταση ανεξαρτησίας με ε, καθόλου πιο εύκολη κατάσταση. Συνεχίζονται οι παλιές διαμάχες, εμποδίζονται η πρόσβαση σε φυσικά ε, κοιτάσματα πετρελαίου και γνωρίζουμε ότι οι παραμεθόριες διαμάχες, ε, οι παραμεθόριες διαμάχες είναι εξίσοξιες ε, και έχουν τραγικές συνέπειες ε, για τον άμαχο πληθυσμό. Με βάση τους εκπροσώπους του ΙΕ και της Ανθρωπιστικής Επιτροπής, πάνω από 500.000 από την περιοχή του Χέγκλικ εκατέλειψαν τις αιστείες τους και οι, περισσότερες, ε, οι περισσότεροι πρόσφυγες έφυγαν ε, ε, από τη χώρα. Έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων. Γιατί λοιπόν δεν αποφύγαμε αυτή την κατάσταση, γιατί πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τις ίδιες καταστάσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είχαμε στην αρχή την εφορία για την ανάκτηση της ανεξαρτησίας και μετά αιματοχυσίες και την εφαρμογή του νόμου του δυνατού. Βέβαια είναι μεγάλο το τίμημα της ε, ελευθερίας, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια λύση στην κατάσταση. Λόγω τώρα στην συνάδελφο κυρία Σάρη Εσαγιά για 1,5 ε, λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα ομόφωνα, ήταν ομόφωνη όταν ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν. Ας μην ξεχνάμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Χαρτούμ. Ε, ε, εκ, εκ μέρους του, από, την πλευρά της είπα ίσως ε, σπεύσαμε να ασχοληθούμε με το χαρτούμ. Τώρα έχουμε μια αποστατικοποιημένη ζώνη η οποία ιδρύθηκε με ένα μηχανισμό ελέγχου και ενέργειες που αναλαμβάνονται ώστε αυτή η αποστατικοποιημένη ζώνη να γίνεται σεβαστή. Πιστεύω ωστόσο ότι θα ήταν χρήσιμο να αρχίσουν και πάλι οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει, διότι αλλιώ θα καταρρεύσει το όλο σύστημα. Πρέπει να προβλέψουμε ένα σωστό καταμερισμό των κοιτασμάτων πετρελαίου. Αυτό που επήγε όμω είναι να λάβουμε υπόψη τη δυστυχία των κατοίκων. Μιλάμε για πάνω από 400.000 άτομα που δεν έχουν καθόλου τρόφιμα. Οι υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών θεωρούν ότι αυτό, ε, κρίνουν ότι αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται διαρκώς εάν συνεχίζει να επιδεινώνεται η κατάσταση και αν παρα... Ε, συνεχίζει η εισρωή τόσων προσφύγων. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Τούνε Κέλαμ για 1,5 λεπτό. Thank you, President. Minister. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι πως μια ε, μακραίωνη σύραξη έχει εξελιχθεί σε ουσιαστική πραγματική διεθνή σύγκρουση που είναι έτοιμη να εκραγεί. Αλλά ομολογώ ότι με ενθαρρύνει ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που ασκούν πίεση στις χώρες αυτές τις καλούν να ακολουθήσουν τον χάρτη πορείας και να καταλήξουν σε μια ειρηνική διευθέτηση. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ενάργεια την, τις κινέζικες, κινέζικες δραστηριότητες γιατί αυτές είναι αποσταθεροποιητικές. Τώρα, ας περάσουμε σε ευχάριστα νέα. Ε, το Συμβούλιο ε, Ασφαλείας ε, θα επεκτείνει κατά έξι περαιτέρω μήνες την παρουσία του στις χώρες αυτές η Ο έλεγχος, ο μηχανισμός ελέγχου οφείλει να αναπτύξει διεθνείς παρατηρητές που θα ελέγχουν επιτόπου τις εξελίξεις. Οφείλουμε βέβαια να εξετάσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση. Περίπου 200.000 πρόσφυγες ε, από το Νότιο Σουδάν επανήλθαν στο Σουδάν μετά την ε, σύγκρουση που προέκυψε. Οφείλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτουν οι βασικές τους ανάγκες για ε, νερό και ιατρική περίθαλψη. Οι τα Ηνωμένα Έθνη μαζί με ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να εμπλακούν σε πιο στρατευμένο χάρτη πορείας. Για 1,5 λεπτό. Κύριε Γκάλα, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ ε, πρέπει να έχει κανεί κατά νου ότι όσον αφορά ε, την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν, με την ανεξαρτητοποίηση αυτή δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Ούτε και όσον αφορά τα τελικά σύνορα. Ο Μάρελ Μπασίρ, ο οποίο έχει την εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ασκεί την εξουσία με τον τρόπο που γνωρίζουμε, ο Μπασίρ λοιπόν ε, εξακολουθεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για πραγματική σταθεροποίηση του Νότου. Υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα διακυβέρνησης στο Νότο και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν με τον τρόπο αυτό θα εμποδίσουμε ε, να υπάρξουν νέες μορφές απεικιοκρατίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει από κοινού. Το ψήφισμα του Συμβουλίου των είναι το πολιτικό και νομικό πλαίσιο. Η δική ευθύνη για την εφαρμογή του ψηφίσματο έχουν εκείνα τα μόνιμα ε, κράτη του Συμβουλίου τη Ευρώπη που έχουν ειδικά συμφέροντα στο χαρτούμ όπω είναι η Ρωσία και η Κίνα. Όλοι ε, πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούμε με την Αφρικανική Ένωση για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Και εγώ πιστεύω ότι οι δυνατόν θα πρέπει να βρίσκουμε αφρικανικέ Λύσει λύσεις για αφρικανικές συγκρούσεις. Σε θέματα πετρελαίου είναι προφανές ότι ο Βορράς και ο Νότος ε, χαρακτηρίζονται από αλληλεξάρτηση. Ο ένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον άλλον. Και όσοι αγοράζουν το πετρέλαιο θα οφείλουν να γνωρίζουν ότι μόνο εφόσον υποβάλλουν ε, στο χαρτούμ και στην Τζούμπα προτάσεις για να τα ξαναβρούν αυτές οι δύο πρωτεύουσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα ε, πρέπει να προχωρήσουν και δεν νομίζω ότι αυτό δεν θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλτών ολοκληρώνεται με τον συνάδελφο κύριο Μπόγκουσλαβ Σόνικ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Μετά το δημοψήφισμα της απόσχεσης ε, και την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν πόρο απέχουν από την εξομάλυση σχέση μεταξύ των δύο χωρών Συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν που στην παραμεθόρια περιοχή βρίσκονται πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ε, επίσης ε, δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη το ύψος των τελών για τη μεταφορά του πετρελαίου, ούτε το νομικό καθεστώς ε, όσων διαμένουν στις παραμεθόριες περιοχές. Ε, και είχαμε ένα δημοψήφισμα το 2011 για την απόσχεση και ε, πραγματικά, επειδή συμμετείχα στην ομάδα παρατήρηση τότε, εκφράζω τεράστια θλίψη μου για την απώλεια ανθρώπινων ζώων, για τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που χρειάστηκε να καταλήψουν τις αιστείε τους και για να σώσουν τη ζωή τους να τραπούν σε φυγή. Δυστυχώς ε, είχαμε ε, πάρα πολλές απώλειες και πολλούς πρόσφυγες. Η διεθνής κοινότητα παρατηρούσε την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ε, ε, και τη δημιουργία νέου κράτους, αλλά ε, δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ο δικός χάρτης για την ειρηνευτική διαδικασία. Δεν καταφέραμε να πείσουμε τις μπλεκόμενες πρεβές για να καθίσουν στο, στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της και στην πράξη και να μην περιοριστεί μόνο σε ωραίε εξαγγελίε που βρίσκονται στα χαρτιά. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye. Ε, δίνω το λόγο στον ε, συνάδελφο κύριο Τάνοκ. The e is deeply concerned about the... Ανασυχούμε πάρα πολύ για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Σουδάν και το το νέο Σουδάν. Εμεί ως ομάδα στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις ε, προσπάθειες ε, του Πρόεδρου σε ε, εξορία να ε, υπάρξουν ε, διαβουλεύσεις ανάμεσα στους δύο νέους πρόεδρους αλλά δεν πρέπει να υπάρξει νέος αιματηρός πόλεμος κυρίως στις περιοχές ε, που αμφισβητούνται όπως το Άμπι και το Χέγκλεκ ο σαφής καθορισμός των συνόρων και ο διαχωρισμός των ενεργειακών αποθεμάτων είναι πρώτη προτεραιότητα στην Τζούμπα δεν υπάρχουν πλέον χρήματα διότι ο αγωγός πετρελαίου έχει κλείσει και η Κίνα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση κατάσταση είναι επικίνδυνη και έχει τρηματίσει όλες τις ελπίδες ε, σχετικά με τις εξελίξεις, ε, την, ε, το διαχωρισμό του Βόρειου από τον Νότιο Σούνταν, ότι δίθεν αυτό θα μπορούσε να επιφέρει κάποια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο είναι ο κύριος Ζέμκε. Ε, unia europejska mm, angażuje się od e, bardzo wielu lat w rozwiązanie konfliktu w sudanie. warto przypomnieć że unia poparła Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με την επίλυση του προβλήματος του ε, Σουδάν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την ανεξαρτητοποίηση του Νοτιού Σουδάν και ε, χορηγεί πολλά εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως αυτή η σύραξη συνεχίζεται. Πρόκειται για μια τραγική σύγκρουση με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Παλαιότερα σε ένα κομμάτι της χώρας υπήρχε η σύγκρουση, τώρα όμως η σύγκρουση αυτή έχει ε, διεθνοποιηθεί και τίθεται ερώτημα κατά πόσον πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κατά πόσον ε, θα πρέπει να έχει τη δική της άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενεργός παίκτη, όμως πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο τα Ηνωμένα Έθνη και η Αφρικανική Ένωση. Ε, οι ομάδες που αναλαμβάνουν διαιτητικό ρόλο ε, πρέπει να είναι από αφρικανικές χώρες. Η κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μία διαμάχη μεταξύ Σουδάν και Ρωτίου Σουδάν θα επηρεάσει την ε, σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τη διεθνή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις δράσεις και τις προσπάθειές της ε, προκειμένου να εφαρμοστεί ο δικός χάρτης στο ΟΗΕ και να εκτονωθεί η κρίση. Χρειάζονται και επιπλέον μέτρα για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μαστίζονται αυτή την ε, πολιτική και οικονομική κρίση. Ο αριθμός των προσφύγων στον καταβλισμό Ίντα έχει διπλασιαστεί μόνο τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στην κατάσταση ε, στην περιοχή Νούμπα. Η Σουδανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει πρόσβαση ούτε καν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Φαίνεται ότι η κρίση είναι τεράστια, δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχουν παιδικές τροφές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ε, πρόσβαση των περιοχών αυτών στη ανθρωπιστική βοήθεια. za vážený pán predsedajúci. Naša podpora vytvorenie novému nezávislého η υποστήριξή μας ε, είναι δεδομένη για το Νέο Σουδάν. Αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουν προκύψει τα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε. Οι διαφωνίες ε, αφορούν τα αποθέματα πετρελαίου στην πόλη Τζούριτς και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μπανκιμούγκ, τις προσπάθειες κατοχής αυτών των ε, περιοχών τις χαρακτήρισε παράνομες. Παρότι λοιπόν το Σουντάν αποσύρθηκε από αυτή την περιοχή, ο πρόεδρος Αμπασίρ απείλησε ε, να κλείσει ο ε, αγωγός. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες για μεταφορά του πετρελαίου, άρα δηλαδή το νότιο Σουντάν εξαρτάται από τη γενοδορία του βόρειου γείτονα. Είναι λοιπόν το ότι δύο χώρες ε, δεν βρίσκονται σε θέση να αναζητήσουν ειρηνευτική λύση και ε, η στρατιωτική σύγκρουση απλά επιτείνει την ε, πείνα. Οφείλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε και τα δύο καθεστώτα ασκούν πίεση. Πρέπει λοιπόν να ξεβρεθεί μία λύση. Είναι ο κύριος Ομπαμάγια. Danke, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το ότι ο Βορράς και ο Νότος ε, συναντιόνται για επίσημες διαβουλεύσεις. Γιατί όπως ξέρουμε η πείνα και η φτώχεια δεν γνωρίζουν ε, σύνορα. Ε, στο Νταφούρ πάψαμε αναστήλαμε την περιουσία μας παρότι ήμασταν εκεί παρόντες για πάρα πολλά χρόνια. Η βοήθεια ε, δεν μπορεί βέβαια να προσφέρεται εις βάρος ε, των ε, κατοίκων στο βορρά. Έχουμε μια μορφή Ισλαμισμού στο νότο αλλά και γενικότερα και στο βορρά έχουμε φιλετικές συγκρούσεις και εκεί αναμειγνύονται χώρες όπως η Κίνα. Αυτά είναι τα αίτια για το ότι αυτή η πολυτάραχη περιοχή δεν μπορεί να ησυχάσει. Η Ευρώπη λοιπόν οφείλει να διαδραματίσει ενεργό σημαντικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο συνάδελφος κύριος Μπρόνς. Μία από τις τραγωδίες ε, στη, στο κέρδος της Δυτικής Αφρικής είναι οι απειλές για εμφύλιο πόλεμο ε, τώρα πια δεν έχουμε φίλιο μόνο πόλεμο στο Σουδάν μετά την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν. Έχουμε μία διαμάχη που είναι η φυσική συνέχεια προηγούμενων συγκρούσεων. Αυτά είναι το κληροδότημα των απεικιοκρατών που χάριζαν τα σύνορα άσχετα με τις εθνοτικές ή τις φιλετικές κοινότητες και έτσι δημιουργήθηκαν συγκρούσεις μετά. Ε, και οι διάφορες φυλές ε, εντός ε, του Σουδάν ε, δεν έχουν μίσχυση μεταξύ τους, άλλοι στο βορρά και άλλοι στο νότο. Επίσης έχουμε δει παρόμοιε περιπτώσεις σε άλλα κράτη που επικρατεί αναρχία. Ε, βέβαια θα πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη γειτονία μεταξύ των δύο τμήματων του Σουδάν. γιατί τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι δύσκολο να διαθετηθούν. Έχουμε ελεύθερη διακίνηση εντό τη Ευρώπη και έχουμε πολλέ φορέ ε, ελεύθερη διακίνηση και υπηκών τρίτων χωρών προ την Ευρώπη. Είναι όμω αυτή καλή ιδέα, αναρωτιέμαι. Στον κύριο Βάμεν Νικολάη, εξ ονόματο τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή και υπάτη εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία. Έχετε το λόγο, κύριε Βάμεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία ως προς τη ε, σοβαρότητα της κατάστασης μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν. Έχουμε ανθρώπινη τραγωδία, τον κόσμο να δεινοπαθεί και έλλειψη πολιτικής βουλής από τις δύο μπλεκόμενες πλευρές για τη διαθέτηση των εκρεμών θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πάρα πολλά για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες που απέφθηναν έκκληση προς το Συμβούλιο να εξακολουθεί να θεωρεί προτεραιότητα του την κατάσταση στο Σουδάν και Νότιο, Νότιο Σουδάν. Εμείς ε, υποστηρίξαμε την διαδικασία ανεξαρτησίας ε, από την ειρηνευτική διάσκεψη του 2005 και στείλαμε δύο αποστολές παρατήρηση εκλογών ε, το 2010 και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν το 2011. Και μάλιστα επικεφαλής των δύο αποστολών ήταν η κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία λοιπόν να ευχαριστήσω και προσωπικά την κυρία Ντεκάιζερ για την στράτευσή της ε, για την περίπτωση του Σουδάν. Και άκουσα τα πολύ σημαντικά σχόλια που είναι καρπός της ε, πλούσιας εμπειρίας που έχετε από την περιοχή. Εμείς υποστηρίζουμε το έργο του πάνελ της Αφρικανικής Ένωσης υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου Τάμπο Μπέκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα ζητά τις εμπλεκόμενες πλευρές να εφαρμόσουν το οδικό χάρτη που προβλέπει το, συμβούλιο του, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ το 2046 και να διευθετήσει τα κρεμή ζητήματα. Ο πρόεδρος του πάνελ Μπέκη είπε ότι θα συγκροτήσει την επόμενη εβδομάδα διάσκεψη στην Αντίσα Μπέμπα, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη. Ευελπιστώντα ότι θα σημειωθεί πρόοδο το συντομότερο δυνατό. σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει τι προσπάθειε τη ε, για την εξασφάλιση Ειρηνη και ασφάλεια στο Σουδάν και Νότιο Σουδάν, ώστε όλοι οι Σουδανοί να μπορέσουν επιτέλου να απολαύσουν του καρπού τη Ειρηνή και τη ασφάλεια. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Βάμεν. κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας με θέμα Γουινέα Μπισάου. Εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και της υπάτης ε, εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας το λόγο έχει ο κύριος Νικολάη Βάμεν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ευτυχής για την ευθερία να συζητήσω σήμερα μαζί σας εξ ονόματος της προσώπου της Αντιπρόεδρου Αύστον την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου. Και χαιρετίζω την